κανονισμό διαπιστώνει το Κοινοβούλιο την χειρία της έδρας του από την 24η Ιουνίου και θα ενημερώνει, ενημερώνει τις εθνικές αρμόδιες εθνικές αρχές. Από